Ich erkläre die διάσκεψη, ε, που διακόπηκε στις 17 Ιουλίου του 2014 επαναλαμβάνεται. Έχω να σας κάνω την ε, λυπηρή